Ρότοβα, Αλεξάνδρ Άλβαρο και τον Σταύρο Λαμπρινίδη για την έλλειψη διαφάνειας και τις ενδυνάμει αντιφάσεις σε σχέση με τη συμφωνία κατά της απομίμησης και προϊόντων μαϊμούδων. Γι' αυτό αυτή η γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού προς όλους τους αποδέκτες διαβιβάζεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής θα καταχωρηθεί εξ ονόματος, με, το όνομα των υπογραψάντων. Και μετά έχουμε και την ε, δήλωση που υποβάλλεται από τον κύριο Ταραμπέλα Κορνέλισεν, Ιλντα Φίγκερέδο και Αντώνια Παρβάνοβα για την διακήρυξη ενός ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Έχει τύχει της ε, υπογραφής της πλειοψηφίας ε, των μελών. Γι' αυτό σύμφωνα με το άρθρο 123 αυτή ε, η δήλωση διαβιβάζεται προς όλους τους αποδέκτες περαιτέρω και καταχωρείται και θα αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας της Ολομέλειας και τα ονόματα των προσυπογραψάντων θα έχουν την αναφορά τους επίσης. Η κυρία Φιγκερέντο έχει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι απλά και μόνο για να ευχαριστήσω, να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ για την υπογραφή όλους τους συναδέλφους που το έκαναν ζητώντας την διακήρυξη, την δημιουργία ενός έτους, ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών θεωρώντας αυτό το θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτή τη δήλωση. Σας ευχαριστώ προς όλους που συνεργάστηκαν. Thank you. ευχαριστώ. Και τώρα, συνάδελφοι, έχουμε επεξηγήσεις ψήφων. Για εκείνους λοιπόν από εσά που δεν θέλουν να επεξηγήσουν την ψήφο τους διαζώσει, α, παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα ώστε να μπορέσουν όσοι επιθυμούν να κάνουν επεξήγηση ψήφου να την κάνουν.